Η μερίσια διάταξη είναι στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να προεδρεύσω τη συνεδριά σα για πρώτη φορά υπό τη νέα μου ιδιότητα. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για την πολύτιμη παρουσία του εδώ και για τα ενδιαφέροντα σχόλια του. Ευχαριστώ τους διερμήνεις και τη δίκηση. Ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλή νύχτα. Και εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση.